and transaction costs and always uh, remaining careful not to increase red tape. Of course the area of freedom, security and justice will bring... Γιατί πιστεύω ότι ούτως ή άλλως ε, θα αναγκαστούμε να υιοθετήσουμε διάφορες νομοθετικές ε, προτάσεις της Κομισιό μέσα στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς, όμως θα πρέπει να, να προσέχουμε έτσι ώστε τι είναι οι νόμοι, αυτές οι νέες προτάσεις να μην ε, επιβάλλουν ε, περισσότερη γραφειοκρατία, περισσότερο κόστος για τις επιχειρήσεις. Ε, εφόσον θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν ενιαίο χώρο, αυτός ο χώρος θα πρέπει να διευκολύνει τους, τους πολίτες, να διευκολύνει τον επιχειρηματικό κόσμο και όχι να δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα. Ευχαριστώ. Ο Κρίστιαν και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος του Όλε Σμιτ, του συναδέλφου μου και μου του ιδίου, θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την τόσο καλά συνδεταγμένη γνωμοδότησή του και φυσικά υποστηρίζουμε την παράγραφο που έχει διατυπώσει. Το πρόγραμμα της Στοχόλμης θέτει τις προτεραιότητες για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας τα επόμενα πέντε χρόνια και η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τα επόμενα χρόνια θα προωθήσει την Ευρώπη των πολιτών και θα εξασφαλίσει ότι οι πολίτες μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και να υποφελθούν πλήρως από την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ο κύριος Σμιτ, ο συνάδελφός μου, έχει κάποιες τροπολογίες, μαζί με αυτόν και εγώ. Θέλουμε καταρχήν να εξασφαλίσουμε την ε, σημασία της αναγνώρισης των επισήμων εγγράφων για να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο αποτελεσματική και κινητική αγορά εργασίας. Επίσης είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε την ε, παραποίηση εγγράφων και προϊόντων και τέλος <clears throat> θέλουμε να παροτρύνουμε τον εισηγητή να μπορέσει να προχωρήσει προς μια ταχύτερη επίλυση των προβλημάτων που συνάπτονται με τις πληρωμές και τις παραδόσεις προϊόντων που αποκτώνται με ηλεκτρονικό εμπόριο διαμεθοριακά. Είναι ένα από τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει. Όσο έχει τώρα η κατάσταση πάντως, Θεωρούμε ότι είναι μια πολύ καλή γνωμοδότηση και είμαι σίγουρος ότι θα έχει μια μεγάλη απήχηση αυτή η γνωμοδότηση και θα υποστηριχθεί γενικότερα. Ευχαριστώ. Δύο ακόμα ομιλητές. Ο Λουί Γκρέκ και η Κάθριν Στάιλερ. Κάποιος άλλος θέλει να λάβει το λόγο. Νομίζω ότι όλοι θα έχουν μιλήσει τότε. Ο Λουί Γκρέκ είναι πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία διευκρίνηση μόνο. Στην γνωμοδότησή σας λέτε ότι ε, προτείνουμε ή συστήνουμε στην Κομισιόν να εντοπίσει τα 20 πιο προβληματικά ε, θέματα. Εγώ πιστεύω ότι η Κομισιόν πρόσφατα έκανε μία προκατακτική ε, πρόταση, ε, δήλωση τέλος πάντων, μια προκαταρκτική δήλωση, το είπε και αυτό ο Επίτροπος η σε απάντηση της επιστολής μου ε, και αναφέρεται επίσης και, στον, και στην χάρτα των πολιτών. Επομένως, οι τροπολογίες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους το γεγονός ότι για αυτά τα θέματα η Κομισιόν ήδη κάτι κάνει. Ναι, καλό θα είναι να αναφερθούμε και στην δική σου έκθεση, να το λάβουμε γι' αυτό υπόψη μας. Σχόλιο εκτός μικροφώνου. Uh, Κύριε Στάιλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θέλω και τον συγγητή. Σύμφωνα με τον προλαλήσαντα τον κύριο Γκρέκ για αυτά τα οποία ανέφερε να αποδώσουμε τα του Κέσαρο στο Κέσαρι όταν κάτι έχει πράγματι γίνει πραγματικότητα. Αυτό είναι σημαντικό να επενέσουμε αυτούς που το πέτυχαν. Θα ήθελα μια διευκρίνηση από τον εισηγητή. Για τα περισσότερα που ανέφερε συμφωνώ απόλυτα. Υπάρχει όμως ένα θέμα το οποίο έχει έρθει στην προσοχή μου. Και έχουμε κάποιες υποθέσεις στα δικαστήρια για το θέμα αυτό. Πρόκειται για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού εντάλματος πώς εφαρμόζεται στην πράξη. Αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι μπορούμε να το εγείρουμε στα πλαίσια αυτής της έκθεσης. Εν γέννη το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης είχε μεγάλη πτυχία στο να φέρει ενώπιον της δικαιοσύνης εγκληματίες που έχουν διαφύγει από τη χώρα όπου έχει διαπραχθεί κάποιο, κάποιο έγκλημα. Αλλά αυτή τη στιγμή η ερμηνεία το ευρωπαϊκό ένταλμα και η ερμηνεία του χρησιμοποιούνται πολλές φορές για ίσονα αδικήματα. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν και κάποια αναθεώρηση ενδεχομένως για να έχει το ευρωπαϊκό ένταλμα την ε, πραγματική σημασία που θα πρέπει να έχει. Νομίζω ότι όλα αυτά τα θέματα είναι χρήσιμο να αντιμετωπιστούν και θα πρέπει να δούμε αν είναι σκόπιμο να εφαρμόζεται αυτό το ευρωπαϊκό ένταλμα σε ίσονους ίσως χαρακτήρα αδικήματα, όπως είπα προηγουμένως. Ευχαριστώ πολύ κυρία Στάιλερ. Μου λέει η γραμματεία ότι τα θέματα αυτά που θίξατε δεν καλύπτονται από την έκθεση της Νομικής Επιτροπής. Είναι μια άλλη έκθεση, αν καταλαβαίνω καλά, μπορεί να με διορθώσει ο κύριος Παντσέρη. Αλλά νομίζω ότι αναφέρεται σε αστικό δίκαιο η έκθεση της Νομικής ε, Επιτροπής, την οποία θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. Εγώ, αν μπορώ να λάβω το λόγο ως σκιώδης, νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό αυτό που λέει η έκθεση, ότι η ενιαία αγορά εδράζεται στη σημαντική αρχή της αμοιβαία αναγνώρισης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε παρακολουθήσει από πολύ κοντά στο πακέτο για τα θέματα των αγαθών και ίσως θα μπορούσε να υπάρχει και κάποια σύνδεση μεταξύ αυτής της, αυτού του πακέτου και της ε, τρέχουσας ε, έκθεσης, γιατί αυτό είναι μία από τις 20 προεξάρχουσες φρούστρες σε ό,τι αφορά τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέρουμε ότι και τα επαγγελματικά προσόντα και αναγνώρισή τους εξακολουθούν να δημιουργούν πολλά προβλήματα. Η κυρία Ρέντινγκ σε μια ομιλία που άκουσα πρόσφατα τόνισε ιδιαίτερα τη σημασία του να εξασφαλίσουμε την αμοιβαία αναγνώριση και εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων σε διαμεθοριακό επίπεδο, ιδίω όταν πρόκειται για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προσπαθούν να ανακτήσουν οφειλόμενα ποσά. Είναι λοιπόν ένα από τα ζητήματα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και είναι ιδιαίτερα καλόδεκτο ότι αναφέρεται αυτό στην εκθεσή σας, στην, στην σας και ότι καταδεικνύουμε στην νομική Επιτροπή ότι αυτό είναι ένα παράγραπτο τμήμα της δημιουργίας της ενιαίας αγοράς και είναι πραγματικά και μια προέκταση, αν θέλετε, αυτών που είπαμε στα πλαίσια της έκθεσης Γκρέκ. Πολύ καλό λοιπόν το περιλαμβάνουμε αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος από την Κομισιόν. Υπάρχει κάποιος από την Κομισιόν που θα ήθελε να σχολιάσει. Όχι. Διακοπές είναι, το ξέρω. Αλλά νομίζω ότι η Κομισιόν θα αντιμετωπίσει εν καιρό την γνωμοδότησή μας. Κύριε Παντσέρη, Νομίζω ότι αναφέρατε το χρονοδιάγραμμα. Ίσως θέλετε να θέλουμε να επανέλθουμε σε αυτό. Οι προθεσμοί για τις τροπολογίες είναι αυτή τη βδομάδα, 30 Σεπτεμβρίου και 29 και 30 Σεπτεμβρίου ψηφίζεται στην Νομική Επιτροπή. Πρέπει όλες οι τροπολογίες να καταδεθούν αυτή τη βδομάδα από τους οικειώδεις και δεν ξέρω κύριε Παντσέρη αν θέλετε να κάνετε κάποια καταληκτικά συμπεράσματα σε σχέση με αυτά που ακούσατε σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιες σύντομες παρατηρήσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την ε, συνεισφορά τους και συνεισφορά που θα υποβάλουν και μέσω των τροπολογιών πιστεύω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε περισσότερο το θέμα το οποίο αφορά την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και ιδίω όσον αφορά την άρση των εμποδίων στην υλοποίηση της ιστορικής αγοράς και ίσως στη συγκεκριμένη περίπτωση να μην ε, αναφερθούμε μόνο σε προθέσεις αλλά να μιλήσουμε και για την ολοκλήρωση ε, της, και της εφαρμογής της οδηγίας ε, για τις υπηρεσίες. Ακούσαμε λοιπόν αυτές τις συστάσεις, θα δούμε τι μπορούμε να προσθέσουμε, με τι θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε. Υπάρχουν δύο απαντήσεις από πλευράς μου. Να αποφύγουμε τη σύραξη με τον Γκρέκ την Ιταλο-Μαλτέζικη και σίγουρα συμφωνώ απόλυτα ότι θα πρέπει αυτή την έκθεσή σου όπως το έκανες να την επανεξετάσουμε και σχετικά με αυτή την πίεση και καταπίεση συμφωνούμε. Θα πρέπει να πούμε ότι τη στιγμή που βλέπουμε ποια είναι τα αρνητικά σημεία που μας ασκούν πίεση να δούμε από πολιτικής πλευράς πώς θα αποφύγουμε την επανάληψή τους. Διαφορετικά τα ίδια θα γίνονται ξανά και ξανά. Συμφωνώ. Ε, καλό είναι να αναφέρουμε λοιπόν, να κάνουμε μια αναφορά και στην εκθεσή σου να αποδώσουμε στον Κέσσαρα αυτό που του ανήκει. Η νομική επιτροπή, κυρίω εκείνη που θα πρέπει να λάβει το λόγο σε αυτονομικά ε, θέματα και στο ένταλμα σε συμφωνώ με τον ε, Πρόεδρο ότι υπάρχουν δύο διαφορετικέ εκθέσεις εδώ. Αναφερόμαστε στον ε, αστικό τομέα, α το πούμε έτσι. Ε, πάντως θα μπορούσαμε να κάνουμε παρόμοια αναφορά προ την κατεύθυνση αυτή γιατί σίγουρα, μα σίγουρα υπάρχει ένα συνδυασμό ανάμεσα στην οικονομική πολιτική εσωτερική αγορά, όπως επίσης και νομικής δικαστικής. Υπάρχει αυτή η σχέση και θα συνεχιστούν τα προβλήματα τα οποία πολύ καλά γνωρίζουμε. Πάντω, επαναλαμβάνουμε, θα μπορούσε να γίνει μια αναφορά όπως είπαμε, όπως είπατε. Αυτά. Σίγουρα θα υπάρξει μια σύγκληση απόψεων, υπάρχει μια σύγκληση απόψεων γύρω από αυτή την έκθεση, είναι κάτι το πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε όπως πρέπει να εφαρμόσουμε αυτό το πρόγραμμα της Στοκόλμης και σας ευχαριστώ. Uh, well, Σας ευχαριστώ πολύ, λέει και ο Πρόεδρος, για την εργασία σας και όλους αυτούς οι οποίοι συνέλαβαν στην ε, επεξεργασία αυτού του θέματος. Κλείνουμε λοιπόν την ημέρησια ατζέντα της συνεδριασής μας. Η επόμενη συνεδρία θα είναι 2 Σεπτεμβρίου. Σας εύχομαι ξεκούραστες και ευχάριστες ε, διακοπές. Να ξαναφορτίσετε τις μπαταρίες σας γιατί έχουμε εντατικό πρόγραμμα του Σεπτεμβρίου. Και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την σκληρά εργαζόμενη γραμματεία μας. Ελπίζουμε ότι θα ξεκουραστείτε κι εσείς. Εκτιμούμε ιδιαίτερα το έργο σας και σας ευχόμαστε και σε εσά καλές διακοπές.